Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Με μεγάλη μου χαρά σας ανακοινώνω την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Εύεν Μάτες ε, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς ε, και την ε, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ χαίρεται που έχει τη δυνατότητα να ακούσει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου μετά από τον πρώτο έλεγχο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός ε, λογοδοτεί στο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και το αρμόδιο μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου έρχεται σε τακτική βάση ε, για ανταλλαγή απόψεων. Πριν μόλις τρεις εβδομάδες η ΕΚΟΝ υπερψήφισε την δεύτερη έκθεση πρωτοβουλίας της που αναφέρεται και στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδιαίτερα όσον αφορά την στελέχωση. Δεν ξέρω αν έχει κάτι να προσθέσεις. Χαιρόμαστε που μπορούμε να παρουσιάσουμε από κοινού την έκθεση αυτή. Ε, δίνω κατευθείαν το λόγο στον ε, κύριο Μάτες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την πρώτη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Γνωρίζετε ε, το πλαίσιο. Ε, η πρωτοβουλία αυτή ε, αποτελέσε αντίδραση στην κρίση και αποφασίστηκε ε, να έχουμε μακροπροληπτική εποπτεία στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Είδαμε μεγάλες ε, διαταραχές ε, στα χρηματοπιστωτικά συστήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μετά από πολλές, πολλά χρόνια ανοχής και υπερβολικής ανάληψης κινδύνου, ε, τελικά έπρεπε οι τράπεζες να βοηθηθούν με χρήματα των φορολογουμένων. Και έτσι δημιουργήθηκε ο ενιαίος αποπτικός μηχανισμός και στόχος ε, ήταν ε, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να υποδεχθεί όλο τον οργανισμό και να έχει και τον γενικότερο έλεγχο. 1.200 οντότητες ελέγχονται και επίσης θα αναλάμβανε ο μηχανισμός την μακροπροεπτική εποπτεία στην Ευρωζώνη γενικά. Ε, προβλέπονταν και πολλέ λειτουργίες. Ε, για παράδειγμα, θα υπήρχε πλήρης αρμοδιότητα όσον αφορά ε, την προστασία του καταναλωτή, τους ελέγχους κατά της νομιμοποίηση παρανομών εσόδων, καθώς και Αυτά είναι πράγματα που διατηρούν τα κράτη-μέλη και επίσης τη μακροπροληπτική εποπτεία. Δεδομένης τη σημασία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, το ελεγκτικό συνέδριο αποφάσισε να ε, κάνει σχετικούς ελέγχους. Ε, καταρχάς, ε, πώς οργανώθηκε ο ενιαίος οπτικός μηχανισμός, πώς οργανώθηκαν οι εργασίες του, ποια είναι η δομή του, πώς, τι ρυθμίσεις λογοδοσίας υπάρχουν και επίσης πώς γίνονται οι επιθεωρήσεις επιτόπου και από μακριά. Τι διαπιστώσαμε λοιπόν. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ότι το σύστημα δημιουργήθηκε σχετικά γρήγορα, μέσα σε 13 μήνες ε, και προσλήφθηκαν ε, περίπου ε, χίλια άτομα. Αυτό ήταν σημαντικό επίτευγμα από μόνο του. Ωστόσο, Διαπιστώσαμε ότι η πολυπλοκότητα του νέου συστήματο αποτελεί πρόκληση και ο νέο μηχανισμό ε, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο συντονισμό και την ε, επικοινωνία ανάμεσα στο προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, και το προσωπικό των κρατών μελών που συμμετέχουν. Επίση, διαπιστώσαμε ότι το Εποπτικό Συμβούλιο δεν έχει έλεγχο του ανθρωπίνου δυναμικού. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του Διευθυντικού Συμβουλίου και επίσης ε, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεσμεύεται από την νομοθεσία να υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στις νομισματικές και τις εποπτικές λειτουργίες του ε, υπάρχουν ε, κάποιες μεικτέ αρμοδιότητες και δεν βρήκαμε να έχουν αντιμετωπιστεί καταλήλως οι σχετικοί κίνδυνοι. Τέλος, ε, διαπιστώσαμε ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ε, ε, προέβλεψε σωστά τις ανάγκες για στελέχωση και έτσι έχει έλλειψη προσωπικού. Επίσης, στις άμεσες επιθεωρήσεις των μεγάλων τραπεζικών ομίλων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη-μέλη. στους 120 μεγάλους ε, ομίλους ε, οι επιτόπου έλεγχοι παίζουν ε, πολύ σημαντικό ρόλο. Μόνο το 20% όμως διευθύνονταν από προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όλοι οι άλλοι έλεγχοι έγιναν με επικεφαλής προσωπικό από τι τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Και δεν υπάρχει μόνο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Επίσης, ε, το εγχειρίδιο για, τους, ε, για την εποπτεία ε, θεσπίζει, καθορίζει ότι θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι με προσωπικό των εθνικών αρμοδίων αρχών. Υπάρχει εδώ μια σύγκρουση ανάμεσα στην πρόθεση των νομοθετών η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ε, ε, επιθεωρεί άμεσα τις μεγάλες τράπεζες ε, και αυτή τη ρύθμιση, ιδιαίτερα τον ρόλο κατά τους επιτόπου ελέγχου των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι γενικά είναι ανεπαρκές το προσωπικό και για τις ομάδες εποπτείας και τις ομάδες ε, επιθεωρήσεων. Αυτό διαπιστώθηκε στην έκθεση. Στο πολύπλοκο αυτό σύστημα έχουμε προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχουμε προσωπικό των ε, Εθνικών Αρμοδίων Αρχών και διαπιστώσαμε σε κάποιο βαθμό ότι το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει σύστημα αξιολόγησης ε, της απόδοσης του προσωπικού που παρέχουν ε, οι εθνικές αρμόδιες αρχές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη, δεν έχει όμως τρόπο να αξιολογεί το προσωπικό που παρέχεται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Επίσης ε, δεν μπορεί να επηρεάσει τις ε, ε, προαγωγές των προσώπων αυτών στις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές, διότι αυτό συγκρούεται με την νομοθεσία κάποιων κρατών μελών. Αυτά λοιπόν ήταν τα βασικά μας ευρήματα. Μπορέσαμε να αξιολογήσουμε την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα κατά τις επιθεωρήσεις επιτόπου και εξ αποστάσεως. Ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμως δεν μοιράστηκε μαζί μας ε, πολλά έγγραφα τα οποία ε, θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητα για τον έλεγχο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεώρησε ότι αυτό ξεπερνάει τα όρια της εντολής μας. Ωστόσο, θεωρήσαμε ότι είναι δικαίωμα του ελεγκτή να αποφασίζει ποια, ποια τεκμηρίωση είναι απαραίτητη για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Πολύ ευχαρίστω θα ακούσουμε την άποψη των νομοθετών πάνω στο θέμα αυτό. Πρέπει να πούμε επίσης ότι η εμπειρία επιβεβαιώνει αυτό που είπαν τα ανώτερα ελεγκτικά όργανα ε, ε, ε, για τον SSM. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν εκάλυψε απόλυτα τις προηγούμενες εθνικές εντολές σε κάποια κράτη-μέλη. Εμείς παρουσιάζουμε και τη διεθνή εμπειρία σχετικά. Θετικά τώρα μιλώντας να πω ότι ε, κάναμε πολλές συστάσεις, ε, περισσότερες από 30 σε 13 ομάδες και η ΕΚΤ δέχτηκε 12. Μία που δεν δέχτηκε πλήρως, εκεί το θέμα αφορά τη δημοσιονομική διαδικασία του προϋπολογισμού, γιατί είδαμε ότι το σύστημα δεν έχει επαρκείς φόρους. Θα πρέπει λοιπόν να ε, υπάρχει μεγαλύτερη εποπτεία και οι ανώτεροι υπάλληλοι, δηλαδή από το Υποπτικό Συμβούλιο, να ε, επηρεάζουν τον προϋπολογισμό. Ε, όμως ε, αναφέρθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, ούτε να υπάρχει υποκλείωση ανθρώπινους πόρους, γιατί δεν είναι ο φορέας λήψης αποφάσεων της έκτα αλλά προστέθηκε από τον κανονισμό για τον εποπτικό μηχανισμό. Οπότε είναι, δε, ε, φτερο, είναι παράγωγη νομοθεσία. Υπάρχει και το θέμα των κοινών υπηρεσιών, των επιμερισμένων, που στηρίζουν και τις δύο λειτουργίες εδώ η έκτη είπε ότι ο πλήρης διαχωρισμός μειώνει την αποτελεσματικότητα, αυξάνει το κόστος. Η σύστασή μας όμως δεν ήταν ότι η χρήση των επιμεριζόμενων υπηρεσιών να εξαλειφθεί τελείως, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος σύγκρουσης στόχων στη νομική υπηρεσία, για παράδειγμα. Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και συστηματικά. Να προσθέσω ότι ε, θεωρούμε ότι η ε, διοίκηση ήταν πολύ επικοδομητική, ε, συνεργάσιμη και μας άκουσε. Άλλωστε είπε ότι δέχτηκε 12 από 13 συστάσεις όπου η μία έγινε μερικώς δεκτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σαμπίνε Λάουτεν Σλέγκαρ αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να σχολιάσω τα αποτελέσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καταρχήν να πω ότι χαιρετίζομαι ιδιαίτερα την εξωτερική προοπτική από το ελεγκτικό συνέδριο σχετικά με το τι βελτιώσεις θα γίνουν σχετικά με την επιχειρηματική ε, λειτουργία, επιχειρησιακή λειτουργία. Υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων γι' αυτό. Η ΕΚΤ συμφωνεί σχεδόν με όλες τις συστάσεις του συνεδρίου και άρχισε δουλειά για να τις εφαρμόσει. Πολλά θέματα ε, έχουμε καταπιαστεί όπως να εξυγχρονίσουμε την διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Έχουμε ένα πλαίσιο ε, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Έχουμε στατιστικές για τις τράπεζες συν νέα επικοινωνιακά μέσα ε, όπως το, ένα φυλάδιο τακτικό ενημερωτικό, ε, αποτελέσματα από workshop, δηλαδή αυξήσαμε τις διαβουλεύσεις με, με, τον κλάδο ε, ακόμα και σε θέματα που δεν χρειάζονται διαβουλεύσεις. Τώρα εξετάζουμε τα προγράμματα δράσης για συγκεκριμένα μέτρα παρακολούθησης, follow-up, ε, μετά τις συστάσεις στην ΕΚΤ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οργάνωση των επιτόπιων επιθεωρήσεων, την εκπαίδευση του προσωπικού, γιατί συμφωνήσαμε για την εκπαίδευση και πώς θα γίνεται στη ε, βελτίωση των συστημάτων πληροφορικής, πληροφοριακών συστημάτων κλπ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις ε, νομικές, τους νομικούς περιορισμούς από το συνομοθέτη. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα, δηλαδή το εύρος της εντολής και αν δώσαμε τα έγγραφα όλα στο ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό ε, θα σας ενδιαφέρει να ακούσετε την άποψή μας. Είμαι πεπισμένος ότι δώσαμε όλα τα στοιχεία ε, για τον έλεγχο που θα ε, πέτρεπε να ασκηθεί η η εντολή του συνεδρίου και να κρυφεί η αποτελεσματικότητα της ΕΚΤ βάσει του άρθρου 27.2 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και το άρθρο 27 του κανονισμού του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Η ΕΚΤ συνεργάστηκε απόλυτα με το συνέδριο για να διευκολύνει τον έλεγχο και έδωσε στην ομάδα του ελέγχου πάρα πολλά σημαντικά έγγραφα, πάνω από 350 και εξηγήσει επίσης που δόθηκαν σε πάρα πολλές συνεδριάσεις στα πλαίσια των ε, νομικών διευθετήσεων που έγιναν. Κάποια έγγραφα, όπως τα πρακτικά του Υποπτικού Συμβουλίου και μεμονωμένες αποφάσεις δεν μπόρεσαν όμως να δοθούν, διότι ο έλεγχος τότε θα ξεπερνούσε την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και θα ε, δημιουργούσε σύγκρουση ε, με την εμπιστευτικότητα σε σχέση με δεδομένα τρίτων. Δεν μιλάμε για πληροφορίες εδώ που έχουμε στη, στα, στις δικές μας βάσεις, αλλά πληροφορίες που έρχονται από τρίτους. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το συνέδριο δεν πήρε πρόσθετες πληροφορίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το συνέδριο ζήτησε ε, διαφορετικές κατηγορίες αποφάσεων σε θέματα κατεπήγοντα, συνήθεις αποφάσεις, ε, ο έλεγχος και αξιολόγηση, για ε, το πρόγραμμα διοδοτήσεων όλη την εσωτερική ροή εγγράφων από την αρχή από την λήψη της απόφασης μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης στη συγκεκριμένη τράπεζα. Και δεν είμαστε σίγουροι γιατί αυτή η συγκεκριμένη τραπεζική τεκμηρίωση χρειαζόταν για να κρυθεί η έκτη και η αποτελεσματικότητά της. Ε, γι' αυτό και για τα θέματα της εμπιστευτικότητας ε, δεν μπορέσαμε να δώσουμε όλη την τεκμηρίωση που περιείχε ε, εμπιστευτικές πληροφορίες για μεμονωμένες τράπεζες. Δώσαμε όμως ένα εξελόφυλλο το οποίο ε, παρουσίαζε ε, αποφάσεις ανωνυμοποιημένες με σύντομη περιγραφή τα διάφορα στάδια της ε, έγκρισης και της απόφασης. Κάναμε δηλαδή ό,τι ήταν δυνατόν για να ε, καλύψουμε το συνέδριο, της ανάγκης του να, στα πλαίσια της εντολής του συνεδρίου που στηρίζεται βέβαια και στην ανεξαρτησία της ΕΚΤ και στις νομικές δεσμεύσεις. Θα ήθελα να πω ότι ο, ο λόγος περιορισμού του εισεντολής ε, αναφέρονται στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης και ο περιορισμός της εντολής του συνεδρίου διασφαλίζει την ανεξαρτησία της έκτο, όπως σας είπα. Ε, ο, κανονισμός ε, SSM χρειαζόταν αλλά θα έπρεπε να ε, συνάδει και να συμμορφούνται προς το πρωτογενές δίκαιο. Ο κανονισμός SSM επίσης δημιουργεί ένα στιβαρό πλαίσιο λογοδοσίας ε, στα πλαίσια του κανονισμού της ΕΚΤΟ, ο κανονισμός SSM, τον SSM και τη διοργανική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μεταξύ άλλων της ε, επανεξετάσεις τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα πρακτικά που στέλνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της Ακροάσης που έγιναν από τον Δανιέλ Λουί σχετικά με την ε, γενικότερη πολιτική και τις επιμέρους τραπεζικές αποφάσεις. Ο, το εύρος της εντολής παράλληλα με το πλαίσιο λογοδοσίας νομίζω ότι διασφαλίζουν ότι αυτό το επίπεδο ελέγχου ε, είναι πολύ θετικός σε σχέση με τα εθνικά πλαίσια. Εμείς ε, ε, είδαμε και την εντολή των εθνικών συνεδρίων και η πλειοψηφία είτε δεν έχει καμία εντολή ελέγχου της εποπτείας ή έχουν πολύ περιορισμένη εντολή, για παράδειγμα τη δημοσιονομική διαχείριση ή την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Από την άποψή μας δηλαδή δεν υπάρχει κενό ελέγχου. Ε, έτσι, ο έλεγχος από την ε, ε, έτσι η ΕΚΤΑ θα, συνεχίσει να είναι ανοιχτή απέναντι στο συνέδριο και θα συνεχίσει ε, τις επικοδομητικές ανταλλαγές με το συνέδριο στα πλαίσια της εντολής του. Και χαιρετίζω ιδιαίτερα τις συστάσεις του συνεδρίου και όπως ε, είπε και ο κύριος Μάτες, με μία μόνο σύσταση δεν συμφωνήσαμε 100% με τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ε, αν αποφασιστεί ποια είδη πληροφορία θα δοθούν από τον ελεγκτή, τότε μπορούν να ανακύψουν προβλήματα. Κύριε Βάλλη, ο εισηγητής, ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για την εργασία αυτή που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και για την Επιτροπή Ελέγχου των προϋπολογισμών και φυσικά θα αποτιμήσουν αυτή την εργασία οι πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα και πιο λεπτομερείς ε, πληροφορίες από την ΕΚΤ, γιατί δεν υπήρχε πλήρης πρόσβαση στις πληροφορίες, γιατί ο εποπτικός μηχανισμός ορίζει ώστε να υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες του ελεγκτικού συνεδρίου για να δοθούν απαντήσεις στους πολίτες. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε γιατί δεν, υπήρχε αυτή η ελεύθερη πρόσβαση όπως θα έπρεπε. Μιλάμε για ένα νέο εποπτικό σύστημα και το σύστημα της ΕΚΤ είναι δεν μπορεί να παραβληθεί με τα εθνικά τραπεζικά συστήματα γιατί δεν είναι ομοιογενή και δεν έχουν τα ίδια τραπεζικά οικονομικά δεδομένα. Η ΕΚΤ λοιπόν δεν έχει τα μέσα για να προβεί σε ένα λεπτομεριακό έλεγχο και στη συνέχεια κρίναμε ότι η εποπτεία δεν ήταν πλήρης και οι εποπτικές αρχές δεν μπόρεσαν να αποτιμήσουν τη διαδικασία ελέγχου. Επίσης, σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο, πολλές φορές ανακύπτουν περιπτώσεις όπου υπάρχει ένας βαθμός αυθαιρεσίας, δηλαδή μία ερμηνεία ανάλογα με τις περιπτώσεις τότε οι εποπτικές αρχές έκριναν ότι δεν μπορούσαν να κρίνουν τα δεδομένα και έτσι τα στοιχεία που είχε η ΕΚΤ από το ελεγκτικό συνέδριο δεν ήταν επαρκή. Επίσης υπάρχει και μία πολιτική σκέψη και ρύθμιση. Δηλαδή στην εποπτεία δεν υπάρχει υπάρχει ένα συστηματικός έλεγχος. Δηλαδή, εμείς δημιουργούμε έναν εποπτικό ε, μηχανισμό και θα πρέπει να δούμε τις αιτίες της κάθε κρίσης. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει υπερβολική χρηματοπιστωτική δραστηριότητα από τις τράπεζες. Ε, δεν λαμβάνονται υπόψη, ας πούμε, παράγοντες όπως η κερδοσκοπία κάτι το οποίο θα έπρεπε να προωθηθεί διαφορετικά. Τι κάνουμε, προβάλλουμε κυρώσεις στον πιστοτικό τομέα, σε μια οικονομία που ήδη νοσεί. Και έτσι δεν προωθούμε την ανάπτυξη και την ανωδική πορεία της Ευρωζώνης. Θα ήθελα να τονίσω, όπως είπε και το ελεγκτικό συνέδριο, ότι η νομισματική πολιτική και ο εποπτικός μηχανισμός, η εποπτεία δηλαδή, γίνονται από το ίδιο όργανο. Άρα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ενδεχομένως. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει μια ανάλυση κινδύνων σε σχέση με αυτές τις επικαλύψεις. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κάτι που έχει απασχολήσει την ΕΚΤ. Δεν ξέρω, και επίσης ε, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ένας διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΚΤ και Ευρωπαϊκού Εποπτικού Μηχανισμού και SSM. Επίσης ε, θα πρέπει ε, να είχαμε ήδη μία πρώτη έκθεση το 2015 για το μηχανισμό SSM. Δυστυχώς όμως ε, δεν δόθηκαν αυτά τα στοιχεία. Άρα η ΕΚΤ δεν δίνει αυτές τις πληροφορίες. Δεν έχουμε ένα πραγματικό δημοκρατικό έλεγχο ως προς τις αποφάσεις της ΕΚΤ. Και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αναλαμβάνει αρμοδιότητες υπερπολαπλάσιες από αυτές που θα έπρεπε και ιδιαίτερα σε, πεδίο, σε περίοδο κρίσης, οι νομισματικές πολιτικές θα πρέπει να αναλαμβάνονται αποκλειστικά από την ΕΚΤ. Ο SSM λοιπόν θα πρέπει να ορίσει τα αίτια των κρίσεων. Ίσως ε, ε, το ότι μιλάμε για τις συνέπειες είναι λανθασμένο. Ίσως φτάσουμε σε ένα πιο ασταθές σύστημα ακριβώς επειδή δεν ορίζονται τα σφάλματα στη βάση. Αυτά ως προς τα σημεία που έθιξε το ελεγκτικό συνέδριο. Και θα ήθελα και οι συνάδελφοι από την ΕΚΟΝ και την ΚΟΝΤ να δώσουν συμπληρωματικές πληροφορίες. Αρχίζουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Χέιες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επικροτήσω αυτήν την έκθεση ε, του ελεκτικού συνεδρίου πάνω στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και επικροτώ και την ε, ε, παρέμβαση του κυρίου Βαλή. Είναι σημαντικό να πούμε ότι ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός δημιουργήθηκε εν μέσω κρίσης ως ο πρώτος πυλώνας μια τραπεζικής ένωσης. Να έχουμε δηλαδή ένα ενιαίο σύστημα εποπτικό, όχι μόνο για τις συστημικά σημαντικές τράπεζες, όπως η Δανιέλα Νόη σε τακτικά χρονικά διαστήματα μα υποβάλλει εκθέσει, αλλά και για τι μη συστημικέ τράπεζε, μικρότερε τράπεζε που υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ ο ενιαίο αποπτικό μηχανισμό δημιουργήθηκε σε μια στιγμή κρίση, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία το Κοινοβούλιο και σε άλλους φορείς. Το ότι το ε, δημιουργήσαμε εν μέσω κρίσης ε, δεν σημαίνει ότι ε, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Πρόκειται για μια μεγάλη οργάνωση με σημαντικό αποτύπωμα στο τραπεζικό μας σύστημα. Και η Δανιέλα Νόη όταν έρχεται στην Επιτροπή μας στην ΕΚΟΝ είναι μία από, τις πιο από τα πιο εξαιρετικά στελέχη και λόγω της γνώσης της, της κατανόησής της ε, και του τρόπου που ε, ε, τα έχει καταφέρει ο ενιαίος αποπτικός μηχανισμός από τότε που δημιουργήθηκε. Και το θέμα δεν είναι μόνο τα stress tests των τραπεζών, το θέμα είναι και το να καθιερώσουμε έναν πολύ σημαντικό δρόμο, έναν πολύ καλό δρόμο για το μέλλον. Και η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου μοιάζει πολύ με την ε, έκθεση ε, που δημοσιεύθηκε πριν ένα χρόνο για το ρόλο της Τρόικας ε, στην διάσωση στην Ιρλανδία. Υπήρχε έλλειψη τεκμηρίωσης, δεν δόθηκαν αρκετά έγγραφα στο ελεκτικό συνέδριο τότε που εξέταζε κάποια θέματα που αφορούσαν την Τρόικα στην Ιρλανδία. Και δυστυχώς ξαναβλέπουμε έλλειψη πλήρους τεκμηρίωσης από πλευράς ε, του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει και θα πρέπει να το τονίσουμε. Δέχομαι ότι έχουν γίνει πολλά. Δέχομαι ότι πολλή δουλειά γίνεται πάνω στο σύστημα ε, της τραπεζικής εποπτείας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βελτιωθεί αυτό και το θέμα της διαφάνειας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ε, βεβαιωθούμε ότι το κοινό καταλαβαίνει την ανάγκη ύπαρξης ε, ενός τέτοιου μηχανισμού. Για μένα είναι απολύτως λογικό, εάν έχουμε ενιαίο νόμισμα και έχουμε και τραπεζική ένωση, να έχουμε και ένα οριζόντιο ευρωπαϊκό σύστημα ε, εποπτικού μηχανισμού. Αυτό όμως θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο σκοπό και θα πρέπει να αποδεικνύει ε, στο κοινό ότι ε, είναι επαρκή τα στοιχεία που δίνει στο κοινοβούλιο και στο κοινό. Θα ήθελα να πω ότι ο, ο διάλογος που έχουμε με τον κύριο Ντράγκη είναι ανεπαρκής. Δεν λαμβάνουμε αρκετές πληροφορίες ε, και χρειαζόμαστε ένα σύστημα με περισσότερη λογοδοσία. Ε, σύντομα λοιπόν ε, για να κλείσω. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να επιτρέπεται να επιλέγει τι έγγραφα θα δώσει στο ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο ε, πρέπει να είναι ο τελευταίος, ο ίστατος φορέας προσφυγής και αποφασίζει εάν ε, ε, ανταποκρίνεται στα πρότυπα ο κάθε οργανισμό ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν μπορεί ε, κάποιο φορέας να πει ότι εμεί απορρίπτουμε την εντολή σα και εμεί αποφασίζουμε τι θα σα δώσουμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την θέση. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό. Ούτε μπορούμε να δεχτούμε, όπω είπε ο συνάδελφο, η έκθεση ανατριετία να μην έχει υποβληθεί ακόμα που θα έπρεπε να είναι ήδη έτοιμη και δέχομαι ότι οι 12 από τις 16 ε, συστάσεις ε, έχουν καλυφθεί. Ε, απλά να κλείσω λέγοντας ότι τα ωφέλη μιας τέτοια έκθεσης είναι ότι μπορούμε να επικεντρωθούμε στις καλές και στις κακές πρακτικές. Χρειαζόμαστε όμως πολύ περισσότερες καλές πρακτικές, ιδιαίτερα με τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιμετωπίζει το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο νομισματικός διάλογος δεν έχει και πολύ σχέση με τον έλεγχο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο νομισματικός διάλογος πάει καλά. Και πολλές φορές το Κοινοβούλιο είπε ότι είναι ικανοποιημένο από το νομισματικό διάλογο και πρέπει να θυμόμαστε και το άρθρο 27.1 και 27.2 της ΕΚΤ ε, αυτό για το περιορισμό του ελέγχου δηλαδή. Υπερβάνος Περέζ. Ναι, υπάρχει διερμηνία, υπάρχει. Είναι πολύ σημαντική αυτή η κοινή συνεδρίαση μεταξύ ΕΚΟΝ και Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εγώ πάντα παρακολουθώ τις εργασίες του ελεγκτικού συνεδρίου και ε, διαβάζω τις εκθέσεις του και θεωρώ ότι και ο μηχανισμός, ο ενίος εποπτικός μηχανισμός και εκπροσωπή θα πρέπει να διαβάσουν τις εκθέσεις αυτές με την ίδια προσοχή. Όμως μεταξύ των νέων θεσμών πολλές φορές δεν λαμβάνεται υπόψη το εύρος της δράσης του SSM. Είναι κάτι που δεν απασχόλησε τόσο πολύ. Δηλαδή μιλάμε για ένα μεγάλο εύρος του τραπεζικού μηχανισμού και τομέα. Και γι' αυτό είναι δύσκολο να επικεντρωθούμε στις μεν ή στις δε πτυχές, γιατί ε, τι κάνουμε, στην ουσία καθιστούμε πιο ε, αδύναμο ένα θεσμό τον οποίο δεν ελέγχουμε τη στιγμή που είναι ο ακρογωνίος λίθος της δράσης μας. Έτσι θα πρέπει να δράσουμε, δηλαδή να συνεισφέρουμε στη διευκόλυνση και στη βελτίωση της εργασίας του SSM. Δεν θα ήθελα να φανώ επικριτική ως προς τον SSM γιατί μιλάμε για έναν πολύ ογκώδη μηχανισμό και δεν θα ήθελα να αφορήσω αυτό το μηχανισμό διότι φυσικά η Τραπεζική Ένωση προτιμούσε σε αρχή φάση να ελέγχει τις εθνικές κεντρικές τράπεζες αλλά τα πράγματα έχουν εξελιχθεί και δεν πρέπει να αποδυναμώνουμε το οικοδόμημα που έχουμε εμείς ε, θεσπίσει. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή εξισορρόπηση με μεταξύ των σφαλμάτων εκκίνησης και της γενικότερης διαχείρισης. Πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος διακατέχεται από επαγγελματικότητα, οι προσλήψεις ε, έγιναν πολύ σωστά, καταρτίστηκε εσωτερικός κανονισμός, οργανόγραμμα και όλα τα σχετικά. Και γι' αυτό νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι λίγο πρόωρη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάλτς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ελεγκτικό συνέδριο, σύμφωνα με, τις κανό... με τους κανόνες, έχει την εντολή να παρακολουθεί την διαχείριση των τραπεζών. Και ως συνομοθέτης εμείς ε, το έχουμε αναθέσει αυτό. Νομίζω ότι πρέπει τους κανόνες ε, και τις συστάσεις του συνεδρίου πρέπει να τις πάρουμε πολύ στα σοβαρά. Όταν μεταφέρονται εθνικές αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά η... ταυτόχρονα δεν ε, μεταφέρεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, ο έλεγχος των λογαριασμών δημιουργείται ένα κενό ελέγχου που πρέπει να κλείσουμε. Η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη ε, και ως ε, υπεύθυνη για την εποπτεία θα πρέπει να φροντίζει για διαφάνεια και να μοιράζεται τις πληροφορίες. Ως Κοινοβούλιο μαζί με την ΕΚΤ στη Διοργανική Συμφωνία ε, σημειώσαμε και αυτό για συγκεκριμένο λόγο ότι οποιαδήποτε μετάθεση εποπτικών αρμοδιοτήτων θα πρέπει να υπόκειται στους κανόνες λογοδοσίας. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να τα τηρεί όλα αυτά. Και η ΕΚΤ ε, δεν πρέπει να ξεχνάει και τον κανονισμό της. Ο κανονισμός λέει ότι η Κεντρική Τράπεζα είναι και νομισματικό όργανο. Ερώτηση προς το συνέδριο. Τι δυνατότητα έχετε να, να, να πείσετε την ΕΚΤ ε, να συνεργάζεται περισσότερο και να έχει περισσότερη διαφάνεια. Και πώς βλέπετε την ιδέα διοργανικής συμφωνίας μεταξύ συνεδρίου και ΕΚΤ. Έχουν γίνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, και μια κυρία, κυρία Λάουντεν Σλέγκελ εδώ, τι λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Τάκουλα παρακαλώ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το, το μέλος, τον κύριο Νέβεν Μάτες για την έκθεση και τον συνάδελφο Μάρκο Μπάλεν για τη συμβουλή, συμβολή τους. Είναι ε, πολύ γρήγορη η σύσταση του SSM στα πλαίσια της ΕΚΤ. Ένα μεγάλο κομμάτι της εποπτείας έφυγε από το εθνικό επίπεδο και πέρασε στην ΕΚΤ. Είναι γι' αυτό πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε στους πολίτες πώς λειτουργεί αυτή η ρύθμιση. Πρέπει να ε, τονίσουμε την ανάγκη πολύ μεγάλη συνεργασίας με το συνέδριο, διαφάνεια μεταξύ των άλλων θεσμικών οργάνων και βέβαια και τα κρατη ε, και η συνεργασία μα, μαζί τους είναι σημαντικά. Συμφωνώ με το συνέδριο ότι θα πρέπει να ε, συμπεριλάβουμε την ε, στην εποπτεία χαμηλότερα επίπεδα, ούτως ώστε να επικεντρωθούμε σε πιο απαιτητικά ζητήματα χρήσιμα για τη λειτουργία του ε, SSM. Ε, αυτό ε, είναι ένα πρόβλημα όταν έχουμε νέες δομές και χρειάζεται χρόνος μέχρι να βρεθεί η τέλεια ισορροπία. Επίσης αναλύεται και η σημασία της συνεχιζόμενης αξιολόγησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγιάλα Σάντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώς ε, δεν μπορεί να είναι παρόν και ο Καταλήν και ζητάει συγνώμη. Έχει να κάνει με την κατάσταση στη χώρα του ή η απουσια του. Θα μου επιτρέψετε όμως να απαντήσω σε κάποιες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο ε, για την ανάλυση της κατάστασης έχει σχολήσει βάθος σε πολλά από αυτά τα θέματα και έχει ασχοληθεί με τις ε, ανησυχίες που ε, έχει εκφράσει ε, και το ελεγκτικό συνέδριο. Έχουμε εδώ λοιπόν μία πρώτη έκθεση για τον μηχανισμό αυτό, αλλά θα συμφωνήσω με την κυρία Περέζ ότι είναι πολύ ε, κρίσιμη στιγμή η παρούσα, είναι ευαίσθητη στιγμή. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τον ε, φορέα αυτόν. Πρέπει να σημειώσουμε ότι έκανε ένα καλό ξεκίνημα και φυσικά είναι σημαντικό να βελτιώνουμε ε, τα πράγματα. Εάν υπάρχουν κάποια προβλήματα ε, ε, τώρα στο ξεκίνημα, θα πρέπει να τα επανορθώσουμε. Ε, θα ήθελα επίσης ε, να πω στον κύριο ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά το ελεκτικό συνέδριο στο πλαίσιο πάντα της κατάστασης. Είναι μια πολύπλοκη και ευαίσθητη η κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Είναι σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε μια έκθεση από τη μία που μπορεί να έχει να κάνει με συγκρούσεις συμφερόντων ή πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, πιθανά προβλήματα, ενδεχομένως συστημικά, αυτό από τη μία και από την άλλη άλλα θέματα που σχετίζονται με τον κίνδυνο. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε την κατάσταση βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να δούμε κατά πόσο αυτά τα firewalls, αυτός ο τείχος αυτά τα τείχη προστασίας υπάρχουν και λειτουργούν έμπρακτα. Θα πρέπει να ορίσουμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία συνεργασίας για να βελτιώσουμε το λειτουργικό πλαίσιο και αυτό κάναμε και μέσα στα πλαίσια της απαλλαγής για το 2015 για να βοηθήσουμε σε θέματα που σχετίζονται με ανθρώπινους πόρους, με περικοπές, γιατί έχει σημασία να δούμε πού ε, βρίσκεται το, το προσωπικό αυτό και πώς δρά. Επίσης η ΕΚΤ θα πρέπει να διαθέσει όλες τις πληροφορίες που επιβάλλονται για έτσι ώστε το ελεγκτικό συνέδριο να μπορεί να υποβοηθηθεί έχοντας στη διάθεσή του όλα τα, τα σχετικά στοιχεία. Έτσι ώστε να υπάρχει μία διαφοροποίηση μεταξύ της εποπτείας υπό την έννοια της επαγρύπνησης και του τραπεζικού εποπτικού μηχανισμού. Είναι βέβαια πολύ λεπτή η διαχωριστική γραμμή γιατί αυτό που μας απασχολεί είναι και η ένταξη των εθνικών κεντρικών τραπεζών σε αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν να ληφθεί υπόψη και αυτό. Γιατί ο καθένας μπορεί να νομίζει ότι ο δικός του τραπεζικός μηχανισμός είναι ο καλύτερος ή δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη από τους άλλους. Να υπάρχει λοιπόν μία εξισορροπημένη προσέγγιση των εθνικών τραπεζικών συστημάτων από την ΕΚΤ και τον SSM. Πέρα από αυτές τις συστάσεις που έχουν μεγάλη σημασία για το μέλλον του συστήματος. Φλάνακαν. Έρχομαι τακτικά στην ε, συνεδρίαση αυτή ε, και όσοι από εσά την παρακολουθείτε συχνά ε, δεν θα εκπλαγούν αυτά που έχω να πω. Πάντα με εντυπωσιάζει ο τρόπος που το ελεκτικό συνέδριο κάνει τη δουλειά του, αλλά όπως είπε και η Πρόεδρος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν επιτρέπεται να επιλέγει τι έγγραφα θα παραδίδει. Νομίζω Πάντω ότι είναι θετική δουλειά που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Και έχω ένα αίτημα. Οι τρει βασικοί στόχοι της Τραπεζικής Ένωσης ε, ε, περιγράφονται εξή εξής. Ε, διαφάνεια, ένωση και περισσότερη ασφάλεια. Ε, ο Ευρωπαϊκός Εποπτικός Μηχανισμός ε, δημιουργήθηκε το 2014 ως ένας από τους τρεις πυλώνες ε, της υποτιθέμενης Τραπεζικής Ένωσης. Τα προβλήματα με το ξεκίνημα στήχησαν 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτοί οι πυλώνες, αυτές οι κολόνες κατέληψαν πάρα τα κεφάλια μας και πριν από το 2014 δεν είχατε λέγει όσον αφορά το τι γινόταν επισήμως, ανεπισήμως όμως ναι. Και ε, είναι χρήσιμο να δούμε ε, τι έγινε στο παρελθόν και να μάθουμε από αυτά ε, όσον αφορά το μέλλον. Στην Ιρλανδία ο Τζόνθαν Σουγκράν πήγε κατευθείαν στο γραφείο του Κεντρικού Ρυθμιστή για τις Τράπεζες και ανακοίνωσε ότι η δική του τράπεζα σε τακτική βάση ε, παραβίαζε τα, τους κανόνες περιρευστότητας και ε, ε, ένα χρόνο μετά όλες οι, τραπεζικές, όλες οι τράπεζες της Ιρλανδίας κατέρευσαν. Κάτι που έκτοτε μας έχει στοιχήσει 17 εκατομμύρια ευρώ. σημαντικά προβλήματα αρχής. Εάν η αρμόδια αρχή είχε ε, εξάγει τότε το λογικό συμπέρασμα ότι αν η μία τράπεζα λέει ψέματα, τότε τι κάνουν και οι άλλες. θα είχαμε λιγότερα προβλήματα. Ακόμα πληρώνουμε όμως 3 ε, ε, δισεκατομμύρια πέρσι, 2 δισεκατομμύρια το προηγούμενο έτος και 1 δισεκατομμύριο το προηγούμενο το πρόβλημα είναι ότι ε, κάψαμε το τραπεζικό μας σύστημα χωρίς να αποφεληθούμε από την ε, ζέστη που ε, δίνει η φωτιά. Δεδομένου ότι η Ιρλανδική Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να αρνείται να αντιδράσει αυτά που είπε ο Τζόναθαν Σούκερμαν, εγώ ρωτά το Ευρωπαϊκό ηλεκτρικό Συνέδριο μήπως ε, θα πρέπει να ελέγχονται, μήπως θα πρέπει να ελεγχθούν οι συνθήκες ε, της υπόθεσης Τζόναθαν ε, Σούκερμαν για να εξεταστούν οι συνέπειες όχι μόνο στον λαό της Ιρλανδίας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Είναι πολύ ακριβά αυτά τα πρώτα προβλήματα, τα προβλήματα των πρώτων δοντιών, όπως λέμε για τα παιδιά. Ε, μπορεί τώρα να λέμε ότι έχει κλείσει η πόρτα, αλλά στο μεταξύ έχει γίνει όλη η καταστροφή. Ε, τώρα πια είναι αργά. Τι, τι μπορεί να κάνει τώρα το ελεκτικό συνέδριο για μας, ε, διότι έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Θέλω να δω τι άλλο μπορείτε να κάνετε. Το λόγο έχει η Γενική Διεύθυνση, η ε, Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση Α, συγγνώμη. Όχι ακόμα. Θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα καταρχήν να κάνω μία δήλωση από πλευράς Γκουε. Εμείς είμαστε υπέρ του δημοσίου ελέγχου του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το θέμα της ε, πίστης είναι πολύ σημαντικό για να το αφήσουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτή είναι η θέση μας καταρχήν. Βεβαίως, σε σχέση με αυτή την απόφαση συγκέντρωσης ε, του ελέγχου, εμείς έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις Το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ SSM και της νομισματικής ε, πολιτικής μέσα στα πλαίσια του ίδιου οργανισμού είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Μία, ένας τέτοιος συγκεντρωτισμός, μία τέτοια συγκέντρωση σημαίνει μέσα τα οποία δεν μπορούμε να προσδώσουμε σε έναν τέτοιο μηχανισμό. Αυτό που χρειάζεται είναι ο συντονισμός μεταξύ SSM και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών για να δοθούν απαντήσεις. Σε σχέση τώρα με τον εποπτικό μηχανισμό βασίζεται στα στοιχεία των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. Θα θέλαμε να ξέρουμε λοιπόν πώς ε, εργάζονται, εργάζεται η υπηρεσία για τη συγκέντρωση αυτών των στοιχείων, διότι ε, κάθε κεντρική τράπεζα έχει ένα δικό της μοντέλο κατάρτισης στοιχείων. Σε σχέση με το shadow banking, και αυτό μας απασχολεί γιατί θα θέλαμε η τράπεζα να είναι υγιής. Αλλά τι κάνει, ε, χρησιμοποιεί την τιτλοποίηση για να ε, εξαγάγει πιστώσεις οι οποίες είναι πολύ ύποπτες. Αυτό το νόημα έχει το shadow banking Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς ορίζονται αυτές οι δράσεις για να αποφευχθεί το shadow banking. Τέλος, σε σχέση με αυτούς τους οργανισμούς too big to fail, αναρωτιέμαι κατά πόσο δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε όχι μόνο με την ε, εποπτεία, αλλά να ασχοληθούμε με τις επενδυτικές τράπεζες και τις ε, ονομαζόμενες λιανικές τράπεζες. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν η Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Όχι, ωραία. Θα ήθελα να δώσω το λόγο για να απαντήσει πρώτα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρακαλώ. Όχι, συγγνώμη, πρώτα στο ελεγκτικό συνέδριο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όσον αφορά το γιατί αναζητήσαμε τα συγκεκριμένα έγγραφα, έχει να κάνει με την εντολή μας. Ελέγχουμε εάν η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εργάζεται αποτελεσματικά. Και γι' αυτό ζητήσαμε τα συγκεκριμένα έγγραφα. Να επιστήσω την προσοχή σας στα αποτελέσματα του ελέγχου μας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχολίασε ότι δεν είναι εντός ε, της εντολής μας. Δεν λάβαμε όμως έγγραφα τα οποία θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητα για τη δουλειά μας. Όσον αφορά ε, τρίτους. Όταν ε, ένας ε, ελεγκτής εξετάζει τα, τους λογαριασμούς σε μιας εταιρείας, είναι φυσιολογικό να ζητάει και στοιχεία άλλων εταιριών, τρίτων. Είναι όμως υποχρεωμένος ο ελεγκτής να σεβαστεί την εμπιστευτικότητα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι στους δημόσιους ελέγχους ε, θα πρέπει να ισχύουν άλλες αρχές. Όσον αφορά το αν μπορούμε να έχουμε κάποια διοργανική συμφωνία, θα πρέπει να πω ότι το Ελεκτικό συνέδριο δεν έχει αποφασίσει ακόμα ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει. Περιμένουμε τα συμπεράσματα του Κοινοβουλίου, καθώς και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν εκδώσει την έκθεσή της για την αναθεώρηση του ενιαίου κοπτικού μηχανισμού. Αλλά αν ακολουθήσουμε αυτή την οδό, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αυτονόητο ότι θα έχουμε επιτυχία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα έτσι. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε να προσπαθήσω καταρχήν να διαλύσω μια παρανόηση. Όλη η πληροφορήση που ήθελε η Κομισιόν σχετικά με τον έλεγχο, αναφέρομαι σε εσά κύριε Βάλη που ρωτήσατε, ότι ήθελαν το δώσαμε. Και οι συνολικές επιχειρήσεις, οι ερωτήσεις, οι ακροάσεις, η τεκμηρίωση, όλα τα προσέφερε, όλα τα παρέσχε η ΕΚΤ. Ε, για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν δική μας η έκθεση ούτε καθυστερήσαμε ε, στην παράδοση κάποιου εγγράφου αλλά αυτό ε, είναι κάποιους μήνες τώρα επίσης εξετάσαμε τα σωστά θέματα όχι μόνο στον πιστοτικό κίνδυνο για παράδειγμα σας διαβεβαιώνω ότι όλα τα, όλους τους κινδύνους τους εξετάζομαι. Κυβερνητική κίνδυνη, κίνδυνη αγοράς, ε, παράγωγα, ε, επίπεδο 3 και κεφαλαϊκή, τιτλοποίηση, ε, επενδυτική τραπεζική, όλα τα κοιτάμε. Σε βάθος, όπως κάνουμε για τον πιστοτικό κίνδυνο. Δεν θέλουμε να αγνοήσουμε κανένα είδος κινδύνου. Εμείς θεωρούμε ότι μόνο οι ανθεκτικές τράπεζες με αρκετά κεφάλαια και αρκετή ρευστότητα με ε, επαρκή διαχείριση κινδύνου, καλά λειτουργική, καλά λειτουργική επιχειρηματική στρατηγική θα μπορέσουν να υπηρετήσουν την πραγματική οικονομία μέσω και μακροπρόθεσμα. Και αυτό περιλαμβάνει την εξέταση του πιστοτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς. Ε, δεν υπάρχει διαφορά εκεί. Και δεν υπάρχει αυθαιρεσία ίσως ό,τι αφορά την εφαρμογή όλων αυτών, γιατί στους ενιαίους κανόνες υπάρχει μεγάλο περιθώριο ε, ελιγμών. Αλλά εμείς ελεγχόμεθα όχι μόνο από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την ε, επιχειρησιακή μας αποτελεσματικότητα, αλλά έχουμε τώρα και την 8 αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να εξετάσει την ικανότητά μας να βλέπουμε επίπεδο 3, παράγωγα κλπ, ε, επιχειρησιακό κίνδυνο. Ε, η Κομισιόν εξετάζει την αποδοτικότητά μας. Έχουμε τον εσωτερικό έλεγχο που τα παρακολουθεί αυτά και υπάρχουν σαφείς κανόνες σχετικά με το, και στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο για το τι είδους αξιολογήσεις πρέπει να κάνουμε. Και είναι σαφές από το ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων ότι πρέπει να διασφαλίσουμε και να έχουμε κατανόηση καλή της επιχειρηματικής στρατηγικής, της στρατηγικής κινδύνου και όλων των κινδύνων στις τράπεζες. Δεν, ε, ε, ε, δεν τιμωρούμε το πιστοτικό κίνδυνο μόνο. Όλα τα κοιτάμε. Για να δούμε τώρα την σύγκρουση συμφερόντων. Έχουμε την αρχή του διαχωρισμού που ε, ε, λειτουργεί στην ΕΚΤΕ και οι κοινέ υπηρεσίες, πληροφοριακό σύστημα, ε, ανθρώπινη πόρη, διοίκηση ε, δεν ασχολούνται με την πολιτική, δεν χαράζουν πολιτική. Την πολιτική τη χαράζει το Εποπτικό Συμβούλιο και το ανώτερο, τα ανώτερα στελέχη του SSM. Και οι μόνοι που είναι στους, και στους δύο τομείς διανόμου αυτό είναι είμαι εγώ που είμαι αντιπρόεδρος του SSM και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και ο, ε, ένα άλλο μέλος. Δεν επηρεάζεται δηλαδή η πολιτική μας και η εποπτεία. Για να δούμε τώρα αν διαλέγουμε αυτά που θα δώσουμε στο ελεκτικό συνέδριο. Σας διαβεβαιώνω και εδώ ότι κάθε αίτημα από το συνέδριο προς εμάς το εξετάσαμε και από νομική άποψη, σε ό,τι αφορά δηλαδή τι υποχρεώσεις απορρέουν από το συνομοθέτη για μας. Είναι σαφές ότι σε κάθε έλεγχο η ενημέρωση από τρίτα μέρη, γιατί όταν κάνετε έλεγχο, κάνετε, κάνετε έλεγχο σε αυτό που πρέπει, σε αυτό που πρέπει να ελέγξετε. Υπάρχει όμως μια σαφής υποχρέωση στον κανονισμό του SSM που λέει επιτρέπεται να δίνουμε πληροφορίες για τράπεζες σε τρίτο μέρος, αν το τρίτο μέρος χρειάζεται να ξέρει. Εδώ ε, περιμένουμε το συνέδριο να κάνει έλεγχο και σε εμά στα πλαίσια της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας, γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει να εξετάζουμε κάθε αίτημα που υποβάλλεται σε εμά να το βλέπουμε και από αυτή την άποψη το κάναμε και για την Κομισιόν. Δηλαδή είδαμε υπάρχει πραγματική ανάγκη να γνωρίζουν. Καμιά φορά, όχι στις περισσότερες περιπτώσεις, το ερώτημα ήταν Δηλαδή γιατί υπάρχει ανάγκη να ξέρετε, γιατί χρειάζεστε για παράδειγμα συγκεκριμένα δεδομένα από μια τράπεζα για να διαπιστώσετε αν η δική μας η διοίκηση είναι αποτελεσματική. Ε, σε δύο λεπτά θα σταματήσει η διαρμηνία, ενημερώνει ο πρόεδρος. Όχι γιατί πρέπει να μιλήσει και ο εισηγητής. Και η τελευταία ερώτηση, πώς δουλεύουμε με τα δεδομένα. Αυτή ήταν, αν θυμάμαι καλά, η τελευταία ερώτηση. Συγκεντρώνουμε τα δεδομένα όλα μαζί, κάνουμε τη συγκριτική αξιολόγηση, το benchmarking και έτσι προσπαθούμε και καταφέρνουμε να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις ε, ε, αυθαιρεσίες, τις αυθαίρετες πληροφορίες. Είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σε ό,τι αφορά την, ε, την συγκριτική αξιολόγηση, την σύγκριση ε, των τραπεζών μας με παρόμοια επιχειρηματικά μοντέλα. Συντομότατα, δύο λεπτά και ο εισηγητής. Με βάση αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση είδα ότι και οι συνάδελφοι συμμετείχαν και έδειξαν ενδιαφέρον το οποίο θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Όλοι μίλησαν για την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας στην ΕΚΤ για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτούς τους μηχανισμούς σε σχέση με απόρριτες πληροφορίες θα πρέπει να φτάσουμε σε μια λύση έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια για την, όπως ακριβώς ζήτησαν και οι πολιτικές ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ για τις αξιολογήσεις σας ως προς το πολιτικό σκέλος. Είδα αποκλήσεις, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν διαφορές που ίσως δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, γιατί όλοι είμαστε Ευρωπαίοι, συμμετέχουμε σε αυτή την ε, Ήπειρο και ε, εάν έχουμε ένα όργανο το οποίο αποδομεί, τότε κανένας δεν ε, αντλεί κάποιο συμφέρον. Γι' αυτό πριν αρχίσουμε της επικρίσεις τη στιγμή που έχουμε το κοινό μας νόμισμα θα πρέπει να κατανοήσουμε αυτές τις αποκλήσεις που υπάρχουν μέσα στα πλαίσια την ΟΝΕ και να εξεύρουμε λύσεις. Μην δημιουργούμε τείχους, μην ε, είμαστε λαϊκιστές, μην επικρίνουμε, ας καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι να βρούμε λύσεις. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να πω ότι ήταν ε, πολύ ανταλλαγή, καλή ανταλλαγή απόψεων. Κατανοώ αυτά που είπε και η ΕΚΤ. Είχαμε πολλές συζητήσεις για τον SSM και θυμάμαι πολύ καλά τι είχαν πει τα μέλη του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού τότε ότι δεν, υπήρχαν, ε, δεν υπήρχαν ανθρώπινοι πόροι. Γι' αυτό νομίζω ότι ε, δεν έχουν εξεταστεί όλα τα επιμέρους ζητήματα. Αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε όταν υπάρχουν προβλήματα, ότι πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Για να αποφύγουμε κινδύνους. Γνωρίζω τους περιορισμούς και των συνθήκων. σε σχέση με την ΕΚΤ και τον SSM ε, τη στιγμή που σε ένα όργανο υπάρχει ένας επιμέρους ε, μηχανισμός και από κοινού. Δεν νομίζω ότι σχετίζεται με τον έλεγχο αυτό. Υπάρχουν θέματα όμως διαφάνειας που θα μας απασχολήσουν λαμβάνοντας υπόψη και την άποψη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους. Εγώ είδα πολύ υποστήριξη για τη θέση του ελεκτικού συνεδρίου. Νομίζω ότι ο κανονισμός ε, ε, ε, για το άρθρο 7, για το άρθρο 2 παραγραφός 7 είναι πολύ σαφής και νομίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε στην έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Λήξη της συνεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και για τη συνεργασία σας.